Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζωζεύ Μανουέλ Παρόζο. Πριν αρχίσουμε όμως την ώρα των ερωτήσεων, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια προς τα πρακτικά. Εάν όχι, εγκρίνονται. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Καλωσορίζω για μία ακόμα φορά τον κύριο Μπαρόζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρχίζουμε με το πρώτο μέρος. Ερωτήσεις από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων και από τα άτομα που ορίστηκαν να υποβάλουν ερωτήσεις εξ των πολιτικών ομάδων. Η ερώτηση ε, για ένα λεπτό και μπορεί να υπάρξει μια επιπρόσθετη ερώτηση 30 δευτερολέπτων και η απάντηση θα πρέπει επίσης να μην ξεπεράσει τα 30 δευτερόλεπτα. Η κυρία Κόρτμαν από το ΕΛΚ έχει το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Βεβαίω, είναι, πολύ... Βεβαίως είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες για την Ευρώπη 2020 για το να υπάρχουν δουλειές πρόοδος και μια καινοτόμος κοινωνική οικονομία της αγοράς. Συγκεκριμένες προτάσεις για